Αφού δεν υπάρχουν ενστάσεις, οι εντολές αυτές επιβεβαιώνονται. Ο κύριος Τσαλίσκι για τις σχέσεις για το Ιράν διορίζεται επικεφαλής γιατί δεν είναι πλέον στην ε, αντιπροσωπεία της Ουκρανίας. Ενστάσεις παρακαλώ. Ε, ορίζεται λοιπόν και αυτή η εντολή. Τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση αν δεν υπάρξουν